ενημερώσω ότι ο κύριος Ζόραν Τάλερ εγκατέλειψε <clears throat> το έδρανό του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την 21η Μαρτίου 2011. Σύμφωνα με τα άρθρα 4 και τα αντίστοιχα άρθρα, σημειώνει το Κοινοβούλιο τη χειρία της ε, θέσης ε, του Ευρωβουλευτού αυτού και θα αναλυθεί η αντίστοιχη δράση αμέσως. Η κυρία Κατρίν Σουλή εγκατέλειψε και εκείνη την θέση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την 24η, από, με σε σχέση με την 24η Μαρτίου θα χειρεύσει η θέση της. Σημειώνουμε την αποχώρηση της ε, κυρίας και θα, θεωρεί, θα θεωρείται ότι θα πρέπει να ε, πληρωθεί η θέση αυτή στο μέλλον. Οι αρμόδιες γαλλικές αρχές ε, με ενημέρωσαν ότι η κυρία Κατρίν Σούλη αντικαταστάθηκε από τον κύριο Μπρίσ Ορτεφέ και μάλιστα από την 24η Μαρτίου 2011. Και στη συνέχεια πιστεύω ότι ο κύριος Όχτεφε βρίσκεται ανάμεσά μας. Κύριε Όχτεφε βρίσκεστε στην Ολομέλεια. Προφανώς όχι. Κυρίες και κύριοι, μια στιγμή, μια στιγμή παρακαλώ. Μάλιστα, το βλέπω, αλλά πρέπει να ολοκληρώσω με τις ανακοινώσεις μου. Μια στιγμή παρακαλώ και σύμφωνα με το κανονισμό 3 όσον αφορά τις διαδικασίες μέχρι ότου θα έχουν ελεγχθεί τα ε, διαπιστευτήρια ε, των ε, μελών που διορίζουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο κύριος Οτεφέ θα μπορεί να παρίσταται στις συνεδριάσεις με τα δικαιώματά του υπό τον όρο ότι προηγούμενα θα έχει υπογράψει μια γραπτή διακήρυξη, μια δήλωση ότι δεν ε, ε, είναι κάτοχος ε, κάποιου άλλου αξιώματος που να είναι ασύμβατο με τη θέση του ως Ευρωβουλευτού. Ο κύριος Κονμπέντιτ παρακαλώ. Ο κύριος Κονμπέντιτ. Κύριε Πρόεδρε, γνωρίζετε τόσο καλά όσο και εγώ ότι υπάρχει μια νόμιμη αντίληψη όσον αφορά τη δυνατότητα του κυρίου Αρτεφέ να γίνει μέλος αυτού του σώματος. Και θεωρώ ότι είναι κάπως απογοητευτικό εκ μέρους της γαλλικής κυβέρνησης να μην περιμένει να επαληθευθεί αυτό. Γιατί ο κύριος Ορτεφέ δεν έχει αποδεχθεί και δεν έχει συμμετάσχει στην ενακτήρια συνεδρίαση του Στρασβούργου και δεν μπορεί συνεπώς να προβεί σε αυτή την αντικατάσταση της κοινή έδρας. Και γι' αυτό ζητώ από το ΕΛΚ ε, να αναμένουν να ληφθεί μια νομική απόφαση για να γνωρίζουμε κατά πόσο ο κύριος Ορτεφέ μπορεί να καταλάβει αυτό το έδρανο. Αλλιώς πρόκειται για ένα σκάνδαλο νομικής ε, φύσεως που έχει ξεσπάσει εδώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Οντί έχει το λόγο όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα και πάλι. Αγαπητέ συνάδελφε, ο κύριος ε, Κον ε, Μπεντίτ ε, δεν, έχει, δεν είναι η πρώτη φορά που δεν δείχνει σεβασμό προς τη δημοκρατία. Ο κύριος Ορτεφέ έχει εκλεγεί αντιπρόσωπο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Ιούνιο του 2009. Αυτό είναι διαφυσβήτητο και ο γαλλικός νόμος το διευκρινίζει. Στην εποχή εκείνη ήταν ε, υπουργός Εσωτερικών και διευκρινίζει ο νόμος ότι ένας υπουργός αυτή τη στιγμή εγκαταλείψει την ε, κυβέρνηση, αποχωρήσει από την κυβέρνηση, μπορεί να καταλάβει αυτή την θέση. Χωρίς μικρόφωνο, δεν ακούγονται οι παρεμβάσεις. Ο Πρίσορτεφέ είχε εκλεγεί αντιπρόσωπο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συμφωνείτε ή όχι. Κοιτάξτε κυρίες και κύριοι, κυρίες και κύριοι. Επιτρέψτε μου να τελειώσω πρόεδρε. Είναι αναφυσβήτητο ότι τα κράτη-μέλη καθορίζουν τους αιρετούς. Ο κύριος Ορτεφέ είχε εκλεγεί, νόμιμα προτάθηκε από τις γαλλικές αρχές να έρχεται και να παίσταται στο κοινοβούλιο. Είναι απαράδεκτα αυτά που ε, αναφέρατε. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Έχω δύο περαιτέρω ανακοινώσει να κάνω. Ε, δύο μάλλον άλλα μέλη ζήτησαν το λόγο. Θα δώσω το λόγο σε δύο συναδέλφους και εκεί θα κλείσει η συζήτηση. Στον πρόεδρο Ντόλ καταρχάς. Θα ήθελα απλώς να πω στο φίλο μου τον κύριο Κονπεντήτ ότι για να μπορεί κανείς να θέσει σε ένα αμφιβόλο μια θέση θα πρέπει καταρχήν να έχει προταθεί. Εάν ε, δεν έχει προταθεί, δεν είναι δυνατόν να αναλύσει η νομική επιτροπή το θέμα αυτό. Λοιπόν, σου προτείνω να κάνεις κάποιους ε, κάποιες προηγούμενες σκέψεις πριν ε, δράσεις, πράτης έτσι ασυλλόγιστα. Ε, είσαι εσύ που μου ζητάς ε, να δείξω σεβασμό προς το δίκαιο. Και τώρα είναι η δική σου σειρά. Θα πρέπει η νομική επιτροπή να αποφανθεί και δεν μπορεί να αποφανθεί παρά μόνο εάν υπάρχει μια επίσημη ε, πρόταση και αν δεν είναι νόμιμη μπορεί η επιτροπή να μας το πει. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκουλάχ έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, εγώ είμαι απόλυτα σύμφωνη με την ιδέα ότι θα πρέπει να περιμένουμε τα αποτελέσματα, τα αποτελέσματα της νομικής ανάλυσης. Θα ήθελα απλώς να πω το εξής, ότι στη δική μας χώρα ε, υπάρχει μια άνοδος ε, των εξτρεμιστών. Και αυτό χωρίς αμφιβολία, επειδή ένα τμήμα της πολιτικής τάξης θεωρούν την εντολή του και τις θέσεις τους ως κάτι το οποίο βρίσκεται αυθαίρετα στη διάθεσή τους. Και από την Γαλλία θα αναμέναμε κάτι περισσότερο. Ιδιαίτερα εφόσον αυτή τη στιγμή στο Κοινοβούλιο έχει την έδρα του στο Στρασβούργο. Σας ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Κυρίε και κύριοι, θα ήθελα για μια στιγμή να επιστρέψουμε στο κείμενο μέχρι ότου επαληθευτούν τα διαπιστευτήρια του μέλους ή έχει ληφθεί απόφαση επιεσδήποτε διαφορά ο κ. Μπρι Οχτεφέ θα πάρει την έδρα του στο Κοινοβούλιο και θα απολαμβάνει όλα τα δικαιώματα τα σχετικά. Υπάρχει μια διαδικασία επαλήθευσης. Πάμε τώρα στα, στην ημερήσια διάταξη. Θα πρέπει να καθορίσουμε την ημερήσια διάταξη για σήμερα και για αύριο το τελικό σχέδιο τη ημερήσια διάταξη που έχει οθετηθεί από, τους, από τη των Προέδρων στις 10 Μαρτίου σύμφωνα με το άρθρο 130 έχει διανεμηθεί και μετά από διαβουλεύσεις πολλές με τις πολιτικές ομάδες προτάθηκε και συμφωνήθηκε να γίνουν